της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικών ε, ζητημάτων για την κατάσταση στις, ε, στη Βενεζουέλα που θα εκπροσωπηθεί από τον κύριο Κούντες. Πριν ξεκινήσει όμως αυτή η συζήτηση θέλω να χαιρετήσω την κυρία Μίτση Καπρίλες Δελεδέσμα η οποία έχει υπήρξε υποψήφιο σε το βραβείο Σαχάροφ το 2015 και την αντιπροσωπεία της από τη Βενεσουέλα που παρακολουθεί τη συζήτηση αυτή ε, για τη Βενεζουέλα από τα διπλωματικά θεωρία. Καλώ ήλθατε. Και τώρα θα δώσω το λόγο και πάλι στον Υπουργό κύριε Κούντες. Ξέρω ότι σε εκπροσωπή κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θέλω να καλωσορίσω και την αντιπροσωπεία από τη Βενεζουέλα. Σας ευχαριστώ που θέσατε το θέμα της Βενεζουέλας στην ημερησία διάταξη. Δύο μήνες μετά από τις εκλογές της 6 Δεκεμβρίου είναι πολύ επίκαιρο το να συζητήσουμε τι αντίκτυπο είχαν αυτές οι εκλογές ή μάλλον δεν είχαν στο πολιτικό και οικονομικό στερέωμα της Βενεζουέλας Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τη συνεχιζόμενη προσοχή που έχει δώσει στην κατάσταση Βενεζουέλα στα τελευταία δύο χρόνια. <clears throat> Από τότε που 43 άτομα ε, έχασαν τη ζωή τους στις βίες ε, ενέργειες που ακολούθησαν διαδηλώσεις ειρηνικές το 2013. Η ενέργειες αυτές έκαναν σαφές ότι η κοινή κρίση αυτή στην Βενεζουέλα μπορεί να ξεπεραστεί μονάχα με επικοδομητικό διάλογο και με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του συντάγματος της Βενεζουέλας. Οι εκλογέ της 6 Δεκεμβρίου είχαν πολύ μεγάλη προσέλευση και οδήγησαν σε αποτελεσμάτα τα οποία ήταν σαφή. Μια σαφής και ισχυρή πλειοψηφία του λαού τη Βενεζουέλα, ζήτησε από το Κοινοβούλιο να πάρει τι απαραίτητε αποφάσει για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσει που αντιμετωπίζει η χώρα. Υποφέρει ο, λαγός, ο λαός της Βενεζουέλας από την κλιμακόμενη, κλιμακούμενη βία. Το Καράκας είναι μια από τις πόλεις με το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρωποκτονιών και απαγωγών στον κόσμο. Οι πολίτες έχουν να αντιμετωπίσουν λήψη βασικών αγαθών, τροφίμων, ε, φαρμάκων και ιατρικής βοήθειας. Με τις εκλογές της 6ης Δεκεμβρίου, ο λαός της Βενεζουέλας ζήτησε να υπάρξει μια πολιτική απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις όλοι οι πολιτικά εμπλεκόμενοι, όλοι οι φορείς πρέπει να σεβαστούν αυτήν την ψηφοφορία για την Εθνοσυνέλευση και επίσης πρέπει να σεβαστούν την ομιμότητα της τωρινής κυβέρνησης. Τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε να βρούμε μια λειτουργική και δίκαια λύση σε αυτά τα προβλήματα. Οι ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, παραθέσεις ή θεσμικές συγκρούσεις δεν θα οδηγήσουν σε καμιά λύση. Δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε, <clears throat> δεν πρέπει να αποδηθούμε σε πολιτικά πολιτικάντικες αντιπαραθέσεις γιατί η οικονομία καταραίει, ο πληθωρισμός γίνεται όλο και πιο έντονος κάθε εβδομάδα. Οι πρωτοβουλίε για ένα εθνικό οικονομικό διάλογο και για μια διαδικασία για να αντιμετωπιστούν τα θέματα των θυμάτων του 2014 έχουν παρουσιαστεί από την εκτελεστική εξουσία. Θα είναι χρήσιμο όλα αυτά αν μπορέσει να υπάρξει μια ανοιχτή διαδικασία με πνεύμα συμβιβασμού και συμφιλίωση. Αυτό απαιτεί σωστό και βαθύ αναλογισμό είναι απαραίτητο να μην ξεχάσουμε την ε, ε, κατάσταση πολλών από τους διαδηλωτές που εξακολουθούν στη φυλακή με αμφισβητήσιμες κατηγορίες. Υπάρχει η περίπτωση του Λεοπόλντο Λόπεθ, ο οποίος ήταν θύμα της βίας που πρέπει να προστατευτεί και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται για βίας ενέργειες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων να τύχουν μιας δίκαιας και ταχείας εκδίκασης της υπόθεσής τους. Όλα αυτά τα θέματα μαζί δημιουργούν μια πολύπλοκη πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί <clears throat> και από τις δύο πλευρές και από την νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία και από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση σε πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού του συντάγματος της Βενεζουέλας. Το Σύνταγμα είναι το μόνο ειρηνικό και νόμιμο πλαίσιο για την πολιτική ζωή της Βενεζουέλας ως αρμόζει σε ένα δημοκρατικό έθνος. Αυτοί που προσπαθούν με παράλληλε δομέ ή με μη συνταγματικέ μεθόδου να αναλάβουν την εξουσία πρέπει να ξέρουν ότι έχουν μια πολύ βαριά ευθύνη. Αν Α είμαστε σαφεί. Αν συνεχίσει η έλλειψη πραγματικού διαλόγου, υπάρχει ο κίνδυνο νέων διαδηλώσεων και βίαιων αντιπαραθέσεων που μπορούν να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο. Ξέρουμε ότι είναι πολλωμένη η κοινωνία της Βενεζουέλας. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο και υπάρχει ένα ιστορικό παρελθόν, αλλά και οι δύο πλευρές θα πρέπει να αποδεχτούν ότι και η άλλη πλευρά έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο. Καμία από τις δύο αντιμεχόμενες πλευρές δεν μπορεί από μόνη να λύσει τα πολλαπλά προβλήματα της Βενεζουέλας. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους φίλους μας στη Βενεζουέλα. Ο διάλογος και ο συμβασμός είναι η μόνη οδός προς τα εμπρός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν αγωνιστεί και στις και το Καράκας θα μεταδώσουν αυτό το μήνυμα και υποστηρίζουμε το μεγάλο αριθμό ε, χωρών εταίρων και περιφερειακών οργανισμών <clears throat> που υποστηρίζουν το διάλογο στη Βενεζουέλα. Η Ευρώπη έχει Θεμητέ ανησυχίε Πάνω από 500.000 πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν στην Βενεζουέλα. Υπάρχουν πολλέ επενδύσει και πολλέ εταιρείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μα απασχολεί και το θέμα τη περιφερειακή σταθερότητα και των δυνητικών αρνητικών αντικτύπων που μπορούν να προέλθουν για τη σύνολη περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στενέ σχέσει με την περιοχή αυτή. συνεργάζομαι, σε πολλά επίπεδα από το εμπόριο ω την ασφάλεια, τον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον αγώνα κατά των ναρκωτικών για να αναφέρω μονάχα μερικέ πτυχέ συνεργασία μα με τη χώρα αυτή. Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τη Βενεσούλα και να την αναβαθμίσουμε. Ξέρουμε ότι πολλοί πολίτες της χώρας αυτής προσβλέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την θεωρούν ένα καλό φύλλο που μπορεί να εξασφαλίσει την διατήρηση του συνταγματικού πλαισίου και της οικονομικής ευμάρειας. Αυτό το έχουμε προσφέρει σε πολλέ από τι θεσμικέ μα συναντήσει στο Καράκα και στι Βρυξέλλε και είναι το μήνυμα που έχω διαδηλώσει δημοσίω σε πολλέ περιπτώσει. Θέλω να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία για να σα ευχαριστήσω για την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για αυτέ τι θέσει και σα ευχαριστώ και για την προσοχή σα. Ευχαριστώ. Θα ζητήσουμε να μιλήσει ο κύριος Γκονζάλες, ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, κάποτε η Βενεζουέλα ήταν ταυτόσιμο με ευημερία και ε, ειρήνη. Ωστόσο, ο τσαβισμός και ο διάδοχός του οδήγησε στην, ε, ερήπο, στα, ε, την Βενεζουέλα στα ερήπια. Δείχνει πως μέσα σε λίγα χρόνια μια χώρα μπορεί να καταστραφεί από την πληστία των ηγετών τους. Αυτό δεν είναι ε, αλλά δεν είναι καταστροφή, είναι κατάρρευση όταν λείπουν φάρμακα και βασικά εργαλεία πρόκειται για μια κατάρρευση του κράτους. Όταν πεινάνε τα παιδιά, όταν στο δρόμο η ζωή του ανθρώπου στοιχίζει λιγότερο από ένα μπιτόνι βενζίνης, πρόκειται για κατάρρευση του κράτους. Όταν άνθρωποι, καλοί, ειρηνικοί φοιτητέ, ε, δημοκρατικοί υποστηρικτές είναι στη φυλακή ενώ οι απαταιώνες είναι στην κυβέρνηση, δεν είναι ε, επανάσταση αυτό, είναι μια κατάρρευση. Ευτυχώ στην Βενεζουέλα φυσάει ο άνεμο του λαού και οι τσαβιστές που προσπάθησαν να βάλουν φυλακή τη δημοκρατία θα δουν ότι η δημοκρατία μπορεί να αλλάξει το καθεστώς δημοκρατικά. Χάρη σε γενναίε γυναίκες όπως η Μίτσι Καπρίλε, η Λίλια Νιμάρη, η Ελευθερία θα βγει από τη φυλακή σε λίγο. Ε, στη Βενεζουέλα. Έλεγε ο Αντώνιο Λεντέσμα ότι δεν διαπραγματευόμαστε την ελευθερία, δεν διαπραγματευόμαστε την δικαιοσύνη, δεν διαπραγματευόμαστε την Βενεζουέλα. Είναι αλήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει ότι με τη Βενεζουέλα πρέπει να είμαστε πάντα στο πλάι του γενναίου λαού τη χώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν δύο κομμάτια στη Βενεζουέλα. Αν υπήρχε, το ένα είναι στην εξουσία, το άλλο είναι στη φυλακή. Ευχαριστώ. Κύριε Γκοντζάλε, υπάρχει μια μπλε κάρτα από την κύριε Σένα Ροντρίγκε. Του δέχεστε? Η κύριε Σένα Ροντρίγκε. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κύριε Πόντ, θα ήθελα να μας εξηγήσετε γιατί στην Γαλλικία ε, στο Ισπανικό κράτος υπάρχουν ακόμα πεινασμένα παιδιά και γιατί στη Γαλλικία υπάρχουν συνδικαλιστές που απειλούνται να φυλακιστούν. Ευχαριστώ. Στη Βενεζουέλα υπάρχει μια φυλακή που λέγεται Λατούμπα. Χτες έναν φοιτητή τον έβαλαν φυλακή χωρίς φυλάκι, χωρίς δίκη, σε, στο πέμπτο υπόγειο, χωρίς φως, χωρίς να έχει επίγνωση που ζει για αόριστο χρόνο και μου λέτε κάτι τέτοια, ντρέπομαι και προτιμώ να μην απαντήσω. Ευχαριστώ. Χαουρέγγι, Ατόντο, δύο λεπτά. Και εγώ θα ήθελα να ε, χαιρετήσω την κυρία Καπρίλες και τους εκπροσώπους και θα ήθελα εξ ονόματος του Κοινοβουλίου να στείλω τρία μηνύματα που θα πρέπει να ακούσει η Βενεζουέλα. Πρώτον, ο λαός της ε, Βενεζουέλα στις 6 Δεκεμβρίου πριν από δύο μήνες μόνο ψήφισε μαζικά. Ψήφισε ειρηνικά και έδωσε ε, την ψήφο του στην αντιπολίτευση. Και το Κοινοβούλιο χαίρεται για αυτή τη δημοκρατική γιορτή και διεκδικεί τη δημοκρατία, γιατί πιστεύει ότι μόνο η δημοκρατία μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα του λαού. Αυτό ήταν το πρώτο μήνυμα. Δεύτερον, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν μπορεί να μειώσει τις εξουσίες της νέας, του νέου κοινοβουλίου που έχει δημιουργηθεί νόμιμα και δεν πρέπει να δημιουργηθούν παράλληλες ε, βουλές, παράλληλα κοινοβούλια για να μειώσουν την νομοθετική εξουσία του πραγματικού Κοινοβουλίου και να δώσουν ξανά μεγαλύτερη εξουσία στην εκτελεστική εξουσία. Γιατί αυτό είναι παραβίαση τη δημοκρατική εντολή που δόθηκε στι 6 Δεκεμβρίου. Τρίτο μήνυμα που θα ήθελα να εκφράσω εν ονόματι πολλών Ευρωβουλευτών. Γιατί υπάρχουν πολλοί που μιλάνε άσχημα για τον Τσάβε. Ε, υπάρχουν άλλοι που τον υπερασπίζονται. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό αλλά και οι δύο ε, απόψεις είναι θεμητές. Θα ήθελα να πω ότι αυτό που είπε πολύ σωστά ο Ολλανδός υπουργό. η λαϊκή εντολή στη Βενεζουέλα είναι μια εντολή διαλόγου ε, για συμφιλίωση. Υπάρχει ένας λαός που θέλει λύσεις. Υπάρχουν δύο ενόμιμες εξουσίες, η εκτελεστική εξουσία και η νομοθετική εξουσία. Και θα πρέπει να συνδιαλλαγούν μεταξύ του. Θα πρέπει να συμφωνήσουν. Γιατί ο λαό θέλει λύσει. Γιατί οι πολίτε θέλουν κανόνε στα τεράστια προβλήματα που υφίσταται η Βενεζουέλα. Έλλειψη ε, εφοδίων, ε, τροφίμων, ε, προβλήματα στην οικονομία. Γι' αυτό θα πρέπει να βρεθούν λύσεις, να, να μιλήσουν για να λύσουν τα προβλήματα για το καλό και το μέλλον της Βενεζουέλας, για το αξίζει ο λαός της. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την ε, κυρία Λεδέσμα που είναι εδώ στα θεωρία και να τους δώσουν υποστήριξη μου. Επίσης τονίζω την ανάγκη να υπάρξει δημοκρατία στην ε, Βενεζουέλα. Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα εγκρίνει τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνει. Εξακολουθούν να υπάρχουν οι δυνάμεις οι οποίες περιστρέφονται γύρω από τον πρόεδρο Μαδούρο και δεν αντιτίθενται στην πλειοψηφία. Είναι απαραίτητο να καταλάβουμε ότι υπήρξε στη Βενεσουέλα μια απόλυτη εξουσία που έχει διαπεράσει όλη την χώρα και αυτή τη στιγμή έχει γεμίσει τις φυλακές με πολιτικούς κρατούμενους. Είναι λοιπόν μια κατάσταση καυχική που επικρατεί στην Βενεζουέλα. Η προσπάθεια πολιτικοποίησης του ανώτατου δικαστηρίου οξύνει ακόμα περισσότερο τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την οικονομική κρίση και τα προβλήματα υγείας στη χώρα. Σε αυτή την τόσο κομική στιγμή η Βενεζουέλα χρειάζεται την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να σε γίνει σεβαστή η αρχή της ε, διάκριση των εξουσιών και του κράτους δικαίου αν δεν προχωρήσει ο νόμος της, ε, της συμφιλίωσης και της αμνηστίας στην Βενεζουέλα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος και για το ίδιο το κράτος δικαίου στην ε, Βενεζουέλα. Ένα λεπτό κύριο Κόουσο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή εδώ και πολλά χρόνια βλέπουμε να γίνονται εκστατείες στη Βενεζουέλα που έχουν σαν στόχο την αποσταθεροποίησή τους. Δυστυχώς πολλοί σε αυτό το ημικύκλιο θέλουν κάτι τέτοιο. Γίνεται σαμποτάζ για τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, επίθεση των μέσων ενημέρωσης, πολιτική βία. 11 νεκροί το 2013, Φεβρουάριο του 2014, μία ε, διαδήλωση με τον Λεοπόντ Λόπες, 44 νεκροί. Στη συνέχεια, πάλι με τον Αντώνιο Λεδέσμο, η επιχείρηση Ιερικό. Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν 20 εκλογικέ διαδικασίες σε 45 χρόνια εξακολουθεί να υπάρχει μια διαδικασία ε, υπονόμευσης του εκλογικού συστήματο. Η αντιπολίτευση θέλησε να κάνει λαθροχειρίες με τις ε, εκλογές του Δεκεμβρίου και ήμουνα ήδη μάρτυρ, μάρτης αυτών. Πάρα πολλοί μίλησαν για εκλογικό ε, πραξικόπημα, αλλά άλλαξαν γνώμη όταν ενίκησαν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση, μια δύναμη η οποία να είναι αν, πάνω από το συνταγματικό σύστημα. Έχουμε ένα πρόεδρο ο έχει την ίδια νομιμότητα όπως οι βουλευτές. Δεν πρέπει εμείς να υποστηρίξουμε τους τομείς αυτούς οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν με τη βία την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Θα πρέπει να διατηρήσουμε την Βενεζουέλα στην κατάσταση μιας δημοκρατίας με αλληλοελεγχόμενες εξουσίες. Υπάρχει μια μπλε κάρτα για σας. Είσαστε έτοιμος να απαντήσετε. Κύριε Κονθάλες Πόνς. Οι τελευταίες εκλογές είχαν διεθνή παρατήρηση. Αυτό το κοινοβούλιο όμως δεν μπόρεσε να πάει γιατί δεν το προσκάλεσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας και δεν μπόρεσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της. Εγώ πήγα εκεί όμως παρόλα αυτά και είδα τι έγινε δεν υπήρξε διεθνής παρακολούθηση. Εγώ ήμουνα παρόν και το ερώτημά μου είναι το εξής. Εσείς πήγατε? Προφανώς ήμουνα. Ακολουθώντας την νομοθεσία της ε, Βενεσουέλας ως παρατηρητής με τον νόμο αυτό που εσείς δεν δέχεστε. Πήγα σε 60 εκλογικά τμήματα, είδα πάρα πολλούς να ψηφίζουν και σε περιοχές της αντιπολίτευσης. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία βία, καμία ε, επιβολή. Όλα αυτά για να καταλάβετε ότι χρησιμοποιείτε ψέματα. Από τον κύριο Φαρία, θέλετε να απαντήσετε το δεύτερο ερώτημα, τη δεύτερη μπλε κάρτα. Κύριε Κόουσο. Όχι. Καλά. Θα συνεχίσουμε τότε. Ο κύριος Σεβαστιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρακαλώ να βάλετε λίγο τάξη στο σώμα που δεν γίνεται, όπου δεν γίνεται σεβασμός ε, κάποιων βασικών κανόνων ε, αυροφροσύνης. Το θέμα είναι η Βενεζουέλα. Ο χρόνος που δίνουμε στην... λίγο από το χρόνο που δίνουμε στη Βενεζουέλα το δίναμε και στο Μεξικό, κοντά γεωγραφικά, μια χώρα με βία, απειλές, ε, επιθέσεις σε δημοσιογράφους. Πρόταση είναι προς τον Υπουργό Νομίζω ότι πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας από τα αποτελέσματα των εκλογών και την διαδικασία την εκλογική, τη δημοκρατική γιορτή που σχολιάστηκε εδώ εκ νέου, διότι και οι προηγούμενες και οι προπροηγούμενες εκλογές είχαν ε, διεθνή υποστήριξη και έγιναν με, δημοκρατικό τρόπο, όπως πάντα. Ποιος είναι ο ρόλος που πρέπει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Βενεζουέλα. Προφανώς να προασπίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί. Αυτό είναι στα, στις συνθήκες. Εγώ ελπίζω να το κάνουμε κάπως καλύτερα από ό,τι το κάναμε σε χώρες όπως το Ισραήλ ή το Μαρόκο, όπου η ατιμορρησία κυριαρχεί και όπου κανείς δεν κάνει τίποτα, αλλά έχουμε πολύ καλές ε, ε, ε, επέσχυντα εγκάδιες θα έλεγα. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε την ειρήνη και για να το κάνουμε αυτό είναι να βοηθήσουμε να αλλάξει αυτό το οικονομικό παραγωγικό μοντέλο που έχει η Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα ανέκαθεν ζει και φοβάμαι ε, ε, ότι οι συνάδελφοι εδώ μιλούσαν για μια ε, εποχή πανέμορφη πριν τον ε, τσαβίσμο που δεν ισχύει. Ζούσε η Βενεζουέλα, ζει πάντα από το πετρέλαιο, κάτι που δημιουργεί αστάθεια, διαφθορά και βία. Αν αυτό που θέλουμε είναι να επαναφέρουμε τις σωστές, τις καλές σχέσεις με την πετρελαϊκή ολιγαρχία για να κερδίσουν οι δικές μας επιχειρήσεις, δεν βοηθάμε το λόγο της Βενεζουέλας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοράο. Ευχαριστώ. Από αυτή την ε, πλεονεκτική θέση μπορούμε να δούμε πώς χρησιμοποιείται η πολιτική για ιδιωτικά συμφέροντα και από τις πολυεθνικές για να αποσταθεροποιήσει ε, και κυβερνήσεις και τη λαϊκή θέληση. Νομίζω ότι υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα στη Βενεζουέλα. Ε, διαφθορά ακόμα και στο κόμμα του Μαδούρο. υπάρχει έλλειψη φαρμάκων, τροφίμων. Υπάρχουν ε, παραστρατιωτικές οργανώσεις. Μπροστά σε αυτή τη την κατάσταση, δυνατές χώρες ή δυνατές περιοχές όπως η Αμερική, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνουν για να βελτιώσουν τη θέση του λαού της Βενεζουέλας. Η απάντηση ε, πρέπει να είναι σαφής. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα οικονομικό πόλεμο απέναντι στην ε, Βενεζουέλα που την κάνει η Τρόικα. Οι επιθέσει προς την ε, Βενεζουέλα τις βλέπουμε όλοι. Ε, κοιτάξτε, κυρώσει από τις Ηνωμένε ε, Πολιτείες που θεωρούν η Βενεζουέλα απειλή για τη χώρα τους. Ε, θα θυμάστε τις ιστερίε κάποιων βουλευτών εδώ μέσα που μιλούσαν για τις εκλογές του Δεκεμβρίου. Εγώ χαίρομαι που ο Μαδούρο δέχτηκε το αποτέλεσμα των εκλογέν και και προσπαθεί να ορθοποδήσει τη Βενεζουέλα. Ευχαριστώ. Ο, Φερ, ο κ. Φερόν. Συνάδελφοι, ευτυχώς δεν συζητάμε μόνο την Ουκρανία. Οι λατινοαμερικανικές χώρες έχουν προορισμό να έχουν προνομιούχες θέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός πολυπολικού κόσμου. Πρέπει να φύγουν από τον θανατηφόρο μαρξισμό. Οι περισσότερες φεύγουν άλλωστε και να αρνηθούν το δόγμα ε, που πριν από δύο αιώνες μετέτρεψε τη Λατινική Αμερική σε, ε, στην πίσω αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών. Η, αυτή τη στιγμή η, οι χώρες, οι παλιές, τα παλιά μαρξιστικά καθεστώτα αντικαθιστούνται από μη μαρξιστικά σε όλες τις χώρες της ε, Λατινικής Αμερικής. Σήμερα ε, το Κοινοβούλιο καλείται να υιοθετήσει και να αποδεχθεί τα αποτελέσματα των εκλογών στη Βενεζουέλα είτε αρέσει είτε όχι στην ΚΟΕ που σήμερα υποστηρίζουν και παλιότερα υποστηρίζαν τις χειρότερες μαξιστικές ε, δικτατορίες. Ο κύριος Μπρόκ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συνεργασία στη χώρα αυτή αλλά δεν υπήρξε αναγνώριση των εκλογών. Έχουν ε, αφαιρεθεί δικαιώματα, έχουν δημιουργηθεί παράλληλα κοινοβούλια. Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης προσπαθούν να δημιουργήσουν μια παράλληλη δομή. Αυτή είναι η θέση εκκίνησης στην οποία βρισκόμαστε. Η Βενεζουέλα είναι μια χώρα από τις πιο πλούσιες χώρες σε πετρέλαιο στον κόσμο και είναι μια από τις πιο φτωχές και με τη μεγαλύτερη εγκληματικότητα στον κόσμο. Όλο και λιγότερο κράτος δικαίου και δημοκρατία παρατηρείται στη δημοσία. Αυτό είναι το σύμβολο του τσαβισμού και του κομμουνιστικού σοσιαλισμού που οδηγεί πάντα σε μεγαλύτερη ένδυα και λιγότερα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι μια εμπειρία που την έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φορές και πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό και με εκπλήτη το γεγονός ότι υπάρχουν βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου όπως ο κύριος Κόουσο που εξακολουθούν να υποστηρίζουν αυτό το σύστημα και να το θεωρούν θετικό. Θα πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε τη θέληση του λαού στην Βενεσουέλα και όχι να προσπαθούμε να την στρεβλώσουμε. Θα ήθελα λοιπόν οι κύριοι του Ποδέμος, οι οποίοι διεκδικούν την συμμετοχή σε κυβέρνηση στην Ευρώπη, να κατανοήσουν ότι η κυβέρνηση μιας χώρας δεν μπορεί να ασκεί τέτοια βία. Ο κύριος Σασί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι υπήρξαν ελεύθερες εκλογές στην Βενεζουέλα. Δεν είναι γεγονός όμως ότι ο πρόεδρος Μαδούρο ανεγνώρισε πλήρως τα εκλογικά αποτελέσματα. Υπήρξε καταρχήν δημιουργία ενός παράλληλου κοινοβουλίου που παραβιάζει τις βασικές αρχές μιας αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Παραβιάζει την αρχή της διάκριση των εξουσιών που είναι η βάση οποιασδήποτε φιλελεύθερης δημοκρατίας. Υπάρχουν αυτέ οι προσπάθειες να στραγγαλίσει την κοινωνία των πολιτών, διατηρώντα πολιτικές προσωπικότητες στη φυλακή μόνο και μόνο επειδή έχουν διαφορετική άποψη με την τωρινή εξουσία <clears throat> στην Βενεσουέλα. Δεν μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο σε μια, δημοκρατικό καθεστώ. Εμεί ω Ευρωπαίοι κοινοβουλευτικοί θα πρέπει να δείξουμε την ε, αλληλεγγύη μας στους βουλευτές που εξελέγησαν μόλις στην Βενεζουέλα. Να τους πούμε ότι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή βρισκόμαστε στο πλευρό τους και θέλουμε να αγωνιστούμε και εμείς ώστε η Βενεζουέλα να ανακτήσει την πολιτική δημοκρατία. Μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλες πτυχές του προβλήματος κοινωνικές και κοινωνικές και οικονομικές, αλλά χωρίς την πολιτική δημοκρατία δεν μπορεί να προχωρήσει μια χώρα. Και αυτό ακριβώς είναι σε διακύβευση αυτή τη στιγμή. Η κυρία Χαράντσοβα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτό που βλέπουμε, νομίζαμε ότι στην Ισπανία θα υπήρχε δημοκρατία, αλλά στην ουσία ο λαός, ε, στον λαό αρνιούνται εξουσίες. Δεν λειτουργεί έτσι η δημοκρατία. Τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Βενεζουέλα. Πρώτον, να επιληθούν τα επίγοντα προβλήματα που επηρεάζουν την οικονομία και την κοινωνία της χώρας. Να υπάρξουν συμφωνίες και όχι συγκρούσεις. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να υπάρξει ένα πραγματικό κλίμα εθνικής συμφιλίωσης. Ποιο το να απελευθερώσουμε όλους τους πολιτικούς κρατούμενους. Δεύτερο, η Ευρώπη πρέπει να είναι περισσότερο παρούσα. Ζητώ από την ύπατη εκπρόσωπο να διευρύνει την εντολή και να αυξήσει τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων μέσων της Ένωσης για να δοθεί απάντηση και να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζει η Βενεζουέλα σήμερα πριν κλείσω να εκφράσω το σεβασμό και τον θαυμασμό μου στις γενναίες γυναίκες της Βενεζουέλας, κάποιες από τις οποίες είναι σήμερα μαζί μας. Τη Μίτσι Καπρίλες, την κόρη της Αντωνιέτα και την Μαρία Αλεχάνδρα Αριστικιέτα, καθώς και την ε, Ταμάρα Σουχού, την Αλίνη Θίαντε τώρα που δεν μπόρεσαν να είναι παρούσε σήμερα. Αυτές είναι ε, μέλη μιας μοναδικής δύναμης για την ελευθερία στη χώρα η αλλαγή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Βενεζουέλα οφείλεται εν πολλής σε αυτές τις γενναίες γυναίκες. Ευχαριστώ. Γκράντες Πασκουάλ, πρόεδρε, η χώρα για την οποία μιλάμε δεν είναι μικρή, ούτε ασήμαντη. Θυμίζω ότι προεδρεύει αυτή τη στιγμή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ το συζητήσαμε το θέμα αυτό και παλιότερα και ζητώντας την ελευθερία ορίσαμε τους πολιτικούς κρατούμενους και η συνάντηση ε, ως υποψήφιος στο βραβείο Ζαχάροφ. Και πήγαμε μόνοι μας γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε μαζί για να δούμε τις εξελίξεις των εκλογών στη Βενεζουέλα. Τι έγινε. Η αντιπολίτευση ανέτρεψε το καθεστώς. Πώς απάντησε όμως το καθεστώς του Μαδούρο. Ε, ε, καθιστώντας ανύπαρκτο το αποτέλεσμα των εκλογών παίζοντας με την εκλογή βουλευτών για να μην υπάρξουν τα δύο τρίτα των βουλευτών τους ώστε να μπορέσει να ανακαλέσουν, να ξεκινήσουν τη διαδικασία ανάκλησης του Προεδρού. Συνεχίζουμε τι κάνουν οι κρατούμενοι, ε, τι κάνουν οι γυναίκες που είναι εδώ. Συνεχίζουν να αγωνίζονται για την ελευθερία και την απελευθέρωση των κρατουμένων που είναι όμως στη φυλακή ακόμα πρέπει να είναι οι φυλακισμένοι, πρέπει να βγουν στο δρόμο και να ασκήσουν πολιτική. Πρέπει να υπάρξει νόμος αμνηστία. Μόνο σε, με, αυτή την προϋπόθεση θα μπορέσει να γίνει διάλογος μεταξύ της κυβέρνησης και της Βουλής, αν θέλει να μιλήσει ο Μαδούρο. Η κυρία Βαλενσιάνο, επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι μερικές ειδήσει, όπως αυτή ότι η δημοκρατία ε, είναι πιο ισχυρή από τις προσπάθειες κάποιων, δεν ισχύει. Μερικές φορές αποδυναμώνεται η δημοκρατία. Νομίζω ότι οι Βενεζουελιάνοι έχουν μπροστά τους ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Ε, μέσω των ε, καλπών μίλησαν, μέσω των εκλογών μίλησαν ε, προέκυψε μια δημοκρατική κυβέρνηση για να γίνουν οι προσπάθειες και οι αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Γιατί χρειάζεται να βγει από μια κατάσταση κρίσης ε, σχεδόν ανθρωπιστική. Δεν θέλω να μιλήσω σαν Ισπανίδα που παίρνει θέση υπέρ του ενός ή του άλλου ε, για τη Βενεζουέλα. Δεν είναι σωστό. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε έκκληση και στην δημοκρατική αξιο... αντιπολίτευση που είναι έχει την πλειοψηφία στον, ε, στο Κοινοβούλιο, καθώς και στον πρόεδρο Μαδούρο, ούτω ώστε να γίνει διάλογος για να ξεκινήσει μια ε, διαδικασία συμφιλίωση στη χώρα. Γιατί αυτό θέλει μέσω των εκλογών ο λαό. Διάλογο, συμφιλίωση, μετάβαση, δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Για μια ακόμα φορά μιλάμε για τη Βενεσουέλα, όπως και στο παρελθόν. Εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως ο Λόπες και ο Λεδέσμα, στη φυλακή όμως. Ο λαός της Βενεζουέλας εξακολουθεί να έχει προβλήματα στην, ε, ε, στην ε, τροφοδοσία με τρόφιμα και ο πληθωρισμός καλπάζει. Είναι η πιο φτωχή και η πιο βίαιη χώρα στην Αμερικανική Ήπειρο. Υπάρχει μια κοινωνική κρίση που εξακολουθεί να μαστίζει τη χώρα αυτή. Αγαπητή κυρία Μίτση, κυρία Αλεξάνδρα, δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Γιατί είναι σαφές ότι είναι η πλειοψηφία των Βενεζολάνων που θέλουν μια αλλαγή για τη χώρα τους και θέλουν να τελειώσει το καθεστώς του Μαδούρο. Φαίνεται όμως ότι ο Μαδούρο δεν δέχεται τη θέληση του λαού της Βενεζουέλας και προσπαθεί να ανατρέψει και να μποϊκοτάρει με κάθε είδους τεχνάσματα τα αποτελέσματα των εκλογών η νέα Εθνοσυνέλευση πρέπει να ζητήσει δημοκρατικές αλλαγές όπως ο νόμος αμνηστίας και συμφιλίωσης για να προωθήσει το σωστό θεσμικό πλαίσιο στην ε, Βενεσουέλα και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ηγηθεί της διεθνούς προσπάθειας να υποστηρίξει αυτή την εθνοσυνέλευση στις μεταρρύθμισεις αυτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να στείλει μια, εθνική, μια επίσημη αντιπροσωπεία για να τονίσει την απερίφραστη υποστήριξή μας στην εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας. Ως Ισπανίδα και ως Ευρωπαία είμαι σίγουρη θα μπορέσουμε να βρεθούμε στο ύψος των περιστάσεων με σαφείς ενέργειες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στίερ. μετά από πολλά χρόνια της αβιστικού καθεστώτος βρίσκεται στα όρια μιας ε, ανθρωπιστικής κρίσης στη Βενεζουέλα. Και αυτό πλήττει κυρίως τα πιο φτωχά στρώματα της κοινωνίας. Είναι μια ανησυχητική κατάσταση και εμείς πρέπει να απαντήσουμε με την αλληλεγγύη μας. Κάντας σαφές όμως ότι αυτή η κατάσταση είναι το άμεσο αποτελέσμα των πολιτικών που έχει ακολουθήσει ένα αυταρχικό καθεστώς το οποίο ξεκίνησε με το να βάλει στη φυλακή όλους τους αντιπολιτευούμενους και αυτή τη στιγμή έχει όμοιρο και στην αθλειότητα όλο το λαό της ε, Βενεζουέλας. Μετά από τις εκλογές της 6ης Δεκεμβρίου εξελέγει μια νέα εθνοσυνέλευση που είναι συμβολική της ανάγκης αλλαγής της κυβέρνησης. Πρέπει ο κ. Ματώνα να αναγνωρίσει τη λαϊκή θέληση, να σταματήσει να προσπαθεί να ελέγξει τη δικαστική εξουσία, να σταματήσει <clears throat> να αναστέλει συνταγματικές ελευθερίες Ζητούμε λοιπόν να υπάρξει αλληλεγγύη με το λαό της Βενεζουέλας, ζητούμε την ελευθερία των πολιτικών κατά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το, ε, το κράτος δικαίου και να φύγει πια το καθεστώς του Τσάβες. Δεν μπορεί ο κύριος Μαδούρο να καταλάβει ότι βυσά νέος άνεμος στη χώρα που γέννησε τον Χωσέ Μαρτί και που από, και ήταν η πατρίδα του Σιμών Πολίβαρο. Ο λαός της Βενεζουέλας ζητά λοιπόν να υπάρξει μια αλλαγή. Πρέπει να είμαστε επάγρυπνοι και να υποστηρίξουμε το λαό της Βενεζουέλας στον αγώνα του για την ελευθερία. Ο κύριος Σουρίνιο έχει το λόγο τώρα. Κύριε Υπουργέ, η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων Ευρώπη και Λατινική Αμερική θα πρέπει να αποτελέσει την προτεραιότητα τη εξωτερική μα πολιτική. Αυτή η προτεραιότητα βασίζεται στην αρχή τη συμπληρωματικότητα των ε, <clears throat> οικονομικών σχέσεων και των αξιών μεταξύ των δύο αυτών πλευρών. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε στην εμπορική συμφωνία με την Σούλ, με την ελπίδα ότι κάποια μέρα και η Βενεζουέλα μπορεί να προσχωρήσει σε αυτή τη συμφωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο όμω δεν μπορούν παρά να τονίσουν την αγανάκτησή του για τι παραβιάσει τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου στην Βενεζουέλα. Η κυβέρνηση Βενεζουέλα θα πρέπει να σεβαστεί το ίδιο το σύνταγμά του Σύνταγμα της χώρας αυτής και τα δικαιώματα των πολιτών και ιδίως των πολιτών και των θεσμών που έχουν εκλεγεί δημοκρατικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τη συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Βενεζουέλα. Αλλά αυτή η συνεργασία πρέπει να έχει και μια κόκκινη γραμμή. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια δικαίου και την ύπαρξη κράτου δικαίου στη Βενεζουέλα. Κύριε Υπουργέ, κυρία ε, Πρόεδρε, πρέπει να τονίσω ότι έχετε όλη την υποστήριξή μας για να ακολουθήσετε σε αυτό το δρόμο για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα. Ευχαριστώ. Μόντ, πρόεδρε, η Δημοκρατική Συμμαχία και η νίκη της ήταν ιστορική νίκη μετά από 17 ε, χρόνια τσαβισμού. Η κατάσταση ωστόσο παραμένει δύσκολη, διότι η απάντηση της κυβέρνησης Μαδούρο δεν ήταν διάλογος, ήταν σύγκρουση Μάλιστα, αλλάζοντας 13 δικαστές του Νότου Δικαστηριού, μειώνοντας τους μηχανισμούς ελέγχου της συνέλευσης, δημιουργεί ενό παράλληλου κοινοτικού κοινοβουλίου ε, από πομπή τριών ε, βουλευτών της ε, νέας πλειοψηφίας. Επιπλέον, ο πρόεδρος διαμορφώνει ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης της κρίσης χωρίς να λάβει υπόψη την, ε, την νικηφόρα αντιπολίτευση την αντίρρηση μεγάλου τμήματος του πληθυσμού και της διεθνούς κοινότητας μεταξύ των οποίων και του Κοινοβουλίου. Και εγώ να καλωσορίσω εδώ την Μίτσι Κατρίλες, υπεύθυνη του Δήμου, την υπεύθυνη του Δήμου ε, του Δήμαρχου, του, τη σύζυγο του Δήμαρχου της Βενεζουέλας. πρόσφατα η πλειοψηφία υιοθέτησε μια πρόταση αποφυλάκησης και αμνηστίας των πολιτικών κρατουμένων που ελπίζουν να ευωδώσει. Αυτό το ζητούσαμε πολλά χρόνια. Η Βενεζουέλα θέλει απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, διάλογο, ανεκτικότητα, συνένεση. Όχι ε, μονομερείς αποφάσεις, κατάχρηση του κράτους δικαίου, απάτη της νομοθεσίας. Μετά από πολλά χρόνια αύξησης του αυταρχισμού και ενός διεθνούς πλαισίου που ε, διευκολύνει την αλλαγή, πρέπει να, να, γίνει, να γίνει αυτή η αλλαγή παρότι συνεχίζει η αντίσταση του καθεστώτος Μαδούρου, ο Σκέλα. Εδώ και 30 χρόνια οι δημοκρατικές εξελίξεις ε, μιας πλούσιας σε φυσικούς πόρους χώρας παραέλυσαν από έντονους ιδεολογικούς πολέμους και αντιπαραθέσεις. Το αποτέλεσμα ήταν το κλασικό. το μοναδικό κόμμα, ε, σοσιαλιστικό κόμμα, επέφερε κοινωνική ε, μιζέρια, ε, διαφθορά, φτώχεια. Πέρυσι η οικονομία συρρυκνώθηκε κατά 10%. Μιλάμε για συγκλονιστικές εξελίξεις. Ακόμα περισσότερο, πριν από δύο χρόνια, 43 πολίτες από της Ανοπλές Δυνάμεις και πάνω από 3.000 ε, συνελήφθησαν. Ο Λεοπόλτο Λόπες μεταξύ αυτών ε, και πολλοί άλλοι είναι ακόμα στη φυλακή. Υπάρχει ένα αίτημα δικαιοσύνης και αλλαγής. Πριν από δύο μήνες εκφράστηκε. Το πρόβλημα είναι ότι ανησυχούμε ότι ο πρόεδρος Μαδούρο δεν είναι έτοιμος να μοιραστεί την εξουσία. Ναι, χρειαζόμαστε εθνικό διάλογο για να ξεπεραστεί η κρίση. Αλλά πάνω απ' όλα η Βενεζουέλα χρειάζεται πραγματικά ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι το κριτήριο για να υπερβούν την κρίση. Ευχαριστώ. Κυρία Χιμένες, θέλετε μπλε κάρτα? Θέλετε να χρησιμοποιήσετε την μπλε κάρτα? Yes. Then... Ποσπισίλ, πρώτος όμως. Πρόεδρε, άκουσα με προσοχή τη συζήτηση και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Συμβούλιο θα πρέπει να ασκήσει απόλυτη πίεση στον πρόεδρο Μαδούρο για να σεβαστεί τα αποτελέσματα των εκλογών. Ωραίο είναι να μιλάμε για διάλογο και συμφιλίωση, αλλά χρειάζονται δύο μέρη για να συζητήσουν. Θα πρέπει και ο πρόεδρος, ο οποίος αυτή τη στιγμή λείπει από το διάλογο. Επίσης, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Δεν μιλάμε για αμνηστία μόνο. Μιλάμε για συνολικές μεταρρυθμίσεις του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα, που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε, τι έκανε το ανώτατο δικαστήριο όταν έδιωξε τρεις ε, βουλευτές. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί η Βενεζουέλα χωρίς ε, δίκαιο και χωρίς ε, σωστό δικαστικό σύστημα. Όλα τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ανησυχητικά και αυτό θα πρέπει να πούμε στη Βενεζουέλα. Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του περασμένου Δεκεμβρίου αποτυπώνει τη δυσαρέσκεια του κόσμου για τη διαχείριση από την προηγούμενη κυβέρνηση της οικονομικής κρίσης που πυροδότησε η ραγδαία πτώση των τιμών του πετρελαίου είναι φυσικό η συγκατοίκηση της νέας κυβέρνησης με τον πρόεδρο μαδούρο να προκαλεί τριβές. το νεοεκλεγέν κοινοβούλιο της βενεζουέλας που κυριαρχείται από την πτέρυγα της αντιπολίτευσης έχει υποσχεθεί να ανατρέψει τις κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης μαδούρο. η αποπομπή τεσσάρων βουλευτών για παρατυπίες κατά την εκλογική διαδικασία συζητήθηκε πολύ στην ευρώπη αλλά δεν είναι το μείζον ζήτημα στη βενεζουέλα σήμερα. άλλωστε ένας εκ των τεσσάρων βουλευτών ανήκει στο κόμμα του κυρίου μαδούρο αντίθετα μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις προκαλεί το νομοσχέδιο που αναμένεται να υπερψηφίσει η νέα βουλή για την ιδιωτικοποίηση των υποδομών κοινωνικής στέγασης σε μια χώρα όπου το 50 του πληθυσμού ζει σε πρόχειρες κατοικίες. απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων της ευρωπαϊκής ένωσης με τη βενεζουέλα με στόχο το αμοιβαίο όφελος των δύο μερών και την τήρηση της αρχής της μη επέμβασης στα εσωτερικά θέματα κάθε μέρους. ευχαριστώ. Κύριος Γιάκοπτσικ. Κύριε Πρόεδρε, οι εκλογές 6 Δεκεμβρίου στη Βενεζουέλα έφεραν ελπίδες στο λαό της Βενεζουέλας. Την ελπίδα ότι θα μπορέσει να υπάρξει ένα μέλλον σε αυτή τη βασανισμένη χώρα που έχει περάσει τόσες μεγάλες δυσκολίες στο παρελθόν και ότι θα μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσουμε τη χρήση των πόρων από, την, ε, από όλο το λαό της Βενεζουέλας και όχι μονάχα από μεμονωμένα άτομα και πολυεθνικές εταιρείε. Πρέπει να τονίσω όμως ότι σήμερα η Βενεζουέλα έχει δύο επιλογές. Ή διάλογος ή χάος. Ή συμφιλίωση ή βία. Αυτοί οι οποίοι θα διαλέξουν την λαθασμένη πλευρά θα είναι υπεύθυνοι για τη συνέχεια στη Βενεζουέλα θέλω να ζητήσω από τους νικητές των εκλογών να δείξουν εγκαρτέρηση και υπομονή να αγωνιστούν για συμφιλίωση και διάλογο και ζητώ και ο ίδιος ο πρόεδρος Μαδούρο να κάνει κάτι τέτοιο αν θέλει το καλό του λαού του. Η κατάσταση σήμερα είναι ε, ξεκάθαρη. Ένας ναρκοδικτάτορος, ο Μαδούρο, κυβερνά τη χώρα και την οδήγησε σε μια ανθρωπιστική κρίση χωρίς προηγούμενο. Επιπλέον, το κοινοβούλιο μας πρέπει να καταγγείλει εκ νέου τα γεγονότα, ζητώντας την απελευθέρωση των άδικα φυλακισμένων πολιτικών κρατουμένων, με διαταγή του Μαδούρο και με την εμπλοκή των ε, δικαστών που είναι ε, ελεγχόμενοι από του Μαδούρο. Ο Μαδούρο είναι ένας καουδίγιο που θέλει να εξαφανίσει όσους δεν συμφωνούν μαζί του. Κυρίες και κύριοι, η καλή Βενεζουέλα, η δημοκρατική Βενεζουέλα που ζητά δημοκρατία και ελευθερία υποφέρει. Είναι αλυσοδεμένη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να ξεκλειδώσει τις αλυσίδες αυτές Ας τολμήσουμε να το κάνουμε και ας απελευθερώσουμε το λαό της Βενεζουέλα. Τελευταίος ο μιλητής, η κυρία Χιμένεθ Μπεκερίλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήμουν μάρτυρας του πώς επετέφθη αυτή η χειρή ε, νίκη της αντιπολίτευσης. Ήμασταν μέσα σε μια μικρή αίθουσα και σας εγγυώμαι ότι η πρώτη κουβέντα που εξέφρασε η αντιπολίτευση ήταν όχι να θριαμβολογήσει κατά του Μαδούρο, αλλά να υψώσουν το χέρι ε, για να χαιρετήσουν τους ε, Βενεζουελιάνους για να υπάρξει ενότητα, θεωρώντας ότι αυτή η ένωση, ε, αυτή η χειρονομία θα την ακολουθούσε και η κυβέρνηση και θα άνοιγε τις φυλακές του, ώστε να βγουν διάφοροι φυλακισμένοι, ο Λεοπόδο Λόπες που είναι μέσα γιατί, γιατί σκέφτονται διαφορετικά, μόνο γιατί θέλουν ελευθερία για τον λαό. Θα ήθελα να χαιρετήσω εδώ την Μίτση Καπρίλες και την κόρη της, τη Μαρία Κολίνα, για διά, διάφορους ε, φυλακισμένους που είναι ακόμα στη φυλακή. Μου είπε μια φυσιοθεραπεύτρια ότι ήταν σε μια ε, διαδήλωση. Θα ήθελα να σας δώσω, να σας χαιρετήσω όλους εσάς και όλο τον Βενεζουελιάνικο λαό δεν πρέπει να κάνετε πίσω. Ακόμα και αν πολλοί εδώ δεν θέλουν να γνωρίσουν ότι δεν υπάρχει οδός πίσω, προς τα πίσω. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινώ λέγοντας ότι είναι σημαντικό να ακούμε τη συζήτηση αυτή και να υπογραμμίσω τη σπουδαιότητα της ε, συζήτησης που είχαμε δύο μήνες μετά τις εκλογές της 6ης ε, Δεκεμβρίου. Η σπουδαιότητα της συζήτησης έγκυται στο ότι οι εκλογές της 6ης ε, Δεκεμβρίου έδωσαν ξεκάθαρα αποτελέσματα. Ο λαός της Βενεζουέλας έδωσε σαφή εντολή στο Κοινοβούλιο για τις αποφάσεις που θα πρέπει να λάβει για να αντιμετωπίσει τις κρίσιμες προκλήσεις της χώρας. Ακούσαμε πολλά για το πώς ως Ευρώπη μπορούμε να βοηθήσουμε στην υλοποίηση μιας διαδικασίας με την οποία θα βγει ο λαός της Βενεζουέλας από την κρίση στην οποία βρίσκεται τώρα. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε την σημασία του συντάγματος. Το σύνταγμα παρέχει ένα νόμιμο ειρηνικό πλαίσιο λειτουργίας της δημοκρατίας της Βενεζουέλας όσοι ένθεν κακήθεν ε, έλκονται από μη δημοκρατικές ε, προσεγγίσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι θα αναλάβουν βαρύτατη ευθύνη σε μια στιγμή που η κατάσταση της χώρας είναι εξαιρετικά σοβαρή οικονομικά και από την οπτική της ασφάλειας. Αν συνεχιστεί η απουσία διαλόγου πρόκειται για ένα κίνδυνο ο κίνδυνος να εκτραχυνθεί η κατάσταση είναι πραγματικός. Ζητούμε λοιπόν να ακολουθηθεί η συνταγματική διαδικασία και να υπάρξει διάλογος. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπογραμμίζουμε κάτι τέτοιο στην πολιτική μας εναντί της Βενεζουέλας. Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε την σπουδαιότητα και εκτιμώ εδώ την παρουσία της αντιπροσωπείας από τη Βενεζουέλα. Ε, είναι σημαντικό έλεγα να δείξουμε ενδιαφέρον και υποστήριξη στην κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό το προωθούμε. Ε, δια, αντλώ από αυτή τη συζήτηση την υποστήριξη στην αντιμετώπιση του, των προβλημάτων της του, του, λαού της Βενεζουέλας και την πολιτική βοήθεια για την υπέρβαση των συγκρούσεων. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να ζητούμε από τους ε, πολιτικούς δρόντες, όλους τους πολιτικούς δρόντες, να ε, επανέλθουν στο διάλογο, σεβόμενοι το Σύνταγμα και, κανείς να μην και να καταλάβουν ότι κανείς δεν μπορεί να δουλέψει μόνος του. Αυτό το κοινοβουλευτικό πλαίσιο που έχετε διαμορφώσει είναι πολύ σημαντικό και ευχαριστώ όσους ταξίδεψαν πέρσι στη Βενεζουέλα για να ακούσουν, να υποστηρίξουν το διάλογο και να υποστηρίξουν το μήνυμα για μια ειρηνική συνταγματική λύση. Είναι πολύ αποτελεσματική όταν υπάρχουν ε, εκπρόσωποι όλων των πολιτικών πλευρών του σώματος, κάτι που ενθαρρύνεται. Εγώ, εμείς ε, ενθαρρύναμε την δυνατότητα να επισκεφθεί η αντιπροσωπεία της τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη χώρα. Να υπογραμμίσω εκ νέου πόσο σημαντικό είναι το ότι το Κοινοβούλιο συνεχίζει να ζητά, να θέτει το θέμα στην ημερήσια διάταξη, ζητώντα την ειρηνευτική διαδικασία στην Βενεζουέλα. Ολοκληρώνεται η σχετική συζήτηση, λέει πρόεδρο. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, η προφορική συζήτηση προ το Συμβούλιο για τη σύμβαση του ΟΗΕ σχετικά με τη διαφορά